votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Για το σχέδιο προϋπολογισμού ε, για το οικονομικό έτος 2011 ε, ο κύριος Φόξ. Ένα λεπτό. Uh, dear, dear colleagues, uh, listen up for a second. We have a lot of explanation. Έχουμε πολλές επεξηγήσεις ψήφου. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με το χρόνο. Θα σας κόβω μετά από ένα λεπτό. Λυπούμε γι' αυτό, αλλά έτσι θα είναι. Εντάξει. Κύριε Φόξ, ένα λεπτό. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να εξηγήσω γιατί Καταψήφισα τον προπολογισμό του 2011. Καταψήφισα γιατί σε περίοδο λιτότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιορίζεται, πρέπει να περιορίζει τις δαπάνες της και όχι να τις αυξάνει. Κατά τη γνώμη μου είναι ντροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αρχικά προτείνει 6% αύξηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με αυτό. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός μου, ο David Κάμερον έκανε καλή δουλειά προσπαθώντας να μειώσει ε, σε 2,9% την αύξηση. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα συμβιβασμό και ο συμβιβασμό αυτό ε, δεν ικανοποιεί ιδιαίτερα του Βρετανού συντηρητικού και ήμουν περήφανος που καταψήφισα την υπερβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία είναι για ένα λεπτό. On merkittävää, että ε, parlamentti ensimmäistä kertaa σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να εγκρίνει τον προπολογισμό και νομίζω ότι στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβλέψει ότι να δώσει μάλλον τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τους δικού τη ιδιού πόρους καθώς επίσης και το τμήμα για το οποίο αποφασίζει αυτή για τον κοινοτικό προπολογισμό και ιδίω όσον αφορά και την περιβαλλοντική πολιτική. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να λάβουμε υπόψη μας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Ευχαριστώ πολύ. Όπω και ο συνάδελφο κύριο Φόξ, συμφωνώ με τι ανησυχίε πολλών Βρετανών συντηρητικών σε περιόδου λιτότητα των κυβερνήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να σφίξουν τα ζωνάρια και να μειώσουν τι ε, δαπάνε του. Πώ μπορούμε να ζητούμε αύξηση που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Είναι η στιγμή που πρέπει να σφίξουμε τα ζωνάρια και να θέσουμε ένα ε, παράδειγμα, να αποτελέσουμε ένα παράδειγμα. Δεν θα έπρεπε να ζητούμε αύξηση ούτε καν ε, διατήρηση του ιδίου επίπεδου. Θα έπρεπε να ζητούμε περικοπές ε, ώστε να πάρουν σοβαρά τους πολιτικούς τους οι φορολογούμενοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ε, τον πόνο τους και προσπαθούμε να τον συμμεριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση Γετζεγεύσκα, η κυρία Ματέρα, για ένα λεπτό. Δεν εδώ. Ο κύριος Γιάρ για ένα λεπτό. Είναι εδώ ο κύριος ε. ε, Είναι το κατεξοχήν δικαίωμα για τον προπολογισμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζει. Ε, χρειάζεται εμπιστοσύνη και εταιρική σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων η διαδικασία των συζητήσεων για τον προπολογισμό του 2011 δεν ήταν μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σεβαστούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι πραγματικά το κατεξοχήν δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήξερα πραγματικά αν βρέθηκα σε κάποια άλλη εποχή τη δεκαετία του 70. Σήμερα δεν ξέρω αν έχω βρεθεί στο 1770. Ο Τόμα Τζέφερσον είχε πει ότι με τέτοια απόσταση οι κυβερνήτες θα πρέπει, μάλλον αναγκαστικά πολλές φορές καταφεύγουν στη διαφθορά και σε κατακριστικές συμπεριφορές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνονται τα ποσά, μόλον ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταβάλει προσπάθειες. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ φορολογίας και εκπροσώπησης. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε να, να επιστρέψουμε τα ποσά αυτά σε αυτά τα οποία ζητεί ε, η κοινή γνώμη είναι να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερη αρμοδιότητα στα εθνικά κοινοβούλια, στους εθνικούς βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται πολύ πιο κοντά στους πολίτες και πρέπει αυτοί να λογοδοτήσουν. Ένα Κύριε Πρόεδρε, Είμαστε υπέρ ε, των μέτρων και ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εποπτεία της ε, ανάπτυξης αυτής της νέας νέου μηχανισμού γιατί υπήρξαν στο παρελθόν ε, πάρα πολλά προβλήματα που είχαν ως αποτέλεσμα ε, κακή ε, οικονομική κατάσταση που με τη συνέχεια της επηρέασε πολλές επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει έλεγχος όλων των αρχών και των κεντρικών τραπεζών ώστε οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοποιητικής ικανότητας να μπορούν να ασκούν το καθήκον τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει τους ελεκτές. Το ποδόσφαιρο οι ε, διαιτητές έχουν ε, διαδικασία έγκρισης και ελέγχου και ό,τι ισχύει για το ποδόσφαιρο θα πρέπει να ισχύει ακόμα περισσότερο για τις κρηματαγορές. Έλεγχος των ελεκτών, των ε, προϊόντων, των οικονομικών, των τραπεζών, ακόμα και κρατών. Αυτό το αναλαμβάνουν οι οργανισμοί ε, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν όμως το έχουν κάνει μονοπόλιο και δεν ελέγχονται οι ίδιοι, τότε γίνονται ιδρύματα που νομίζουν ότι είναι θεοί και πάμε και τους οικετεύουμε. Δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα, το λένε και οι δέκα ειδωλές, να μην λατρεύεις άλλο Θεό εκτός από μένα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, διορθωθεί αυτή η στρέβλωση με αυτή την έκθεση και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξαναρωτήσει και να ξαναζητήσει να δει αν έχουν γίνει όλα αυτά πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Έκθεση για κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίσαμε για τον προπολογισμό του 2011 και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ξεκινάει μια νέα διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη αλλά τουλάχιστον μας δίνει κάποιες νέες αρμοδιότητες. Κάναμε κάποιους συμβασμούς, έκανε κάποιες θυσίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο. Καταφέραμε όμως παρόλα αυτά να θέσουμε παραμέρος τον κίνδυνο του 12 τιμωρίου, το οποίο θα είχε πολύ δυσχερείς επιπτώσεις για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε όμως να δούμε ακριβώς ποιοι είναι υπεύθυνοι για την αποτυχία του προγράμματος ΙΤΕΡ, καθώς επίσης και για το ζήτημα της ευελιξίας. Έχασε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους διεθνείς εταίρους. Δεν θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια σημαντικά κοινοτικά προγράμματα δεν θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε δραστηριότητες οι οποίες απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες, αλλά είμαστε και σε θέση να τις χρηματοδοτήσουμε για το μέλλον. Το πήρα από το ρελέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ανάγκη εξυγχρονισμού της ε, μετρολογίας των σταθμών που χρησιμοποιούμε, όπως επίσης και βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας, μας ε, οδηγεί στην εφαρμογή της οδηγίας για τη μετρολογία. Είναι το πρώτο, το πρώτο βήμα για να υπάρξει μια πιο συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ε, επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Είναι επίσης ε, σημαντικό να αποφασίσουμε ποιες πρέπει να είναι οι προθεσμίες ε, για να μπορέσει να αξιολογηθεί από τα κράτη-μέλη του αντικτύπου της κατάργησης σχετικής νομοθεσίας και για να μπορέσουμε να διορθώσουμε ορισμένα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουμε. Η επιλογή των ε, εξαιρέσεων ε, είναι πολύ σωστή στο πλαίσιο των οδηγιών αυτών ε, και στο πλαίσιο μεγαλύτερη απλοποίηση. Ελπίζουμε όμως να μην χειροτερέψουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόντε για ένα λεπτό. Ρόντε. No. Ο κύριος Μαστέλα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει βασική καινοτομία στη λειτουργία, τη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η πρωτοβουλία των πολιτών όντως εισάγει ένα νέο ε, σύστημα διεθνικής ε, δημοκρατίας και συμμετοχικής μάλιστα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορέσουν λοιπόν όλοι οι πολίτες ε, να απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα και υποστηρίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη δεχόμαστε ευνοϊκά, τη συμμετοχή της των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών είναι σημαντική και ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων μας και την ένωση στα μάτια των πολιτών της. Η κυρία Μπιλμπάο, για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ. Ε, ο κύριος Γιουνκέρας για ένα λεπτό. Gracias, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση τη ε, πρωτοβουλία πολιτών. ο σκιώδη ηγητή στην Επιτροπή Πολιτισμού και λυπάμαι όμω που δεν εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο δύο ζητήματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, το ότι ε, οι νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να είναι και αυτοί σε θέση να υπογράφουν, να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και η ψήφωση στη συνέχεια των Προέδρων δεν εγκρίθηκαν τα δύο αυτά σημεία και γι' αυτό το λόγο και εμείς αντιταχθήκαμε και καταψηφίσαμε σε αυτά συγκεκριμένα αυτά σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόντε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ψήφισα υπέρ της πρωτοβολίας των πολιτών για να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πιο κοντά τους η Ένωση. Τώρα έχουμε μια ομοιόμορφη διαδικασία ε, για όλα τα κράτη-μέλη για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και θέλουμε να είναι ένα εύχριστο εργαλείο. Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να προέρχονται από το 1 τέταρτο των κρατών μελών τουλάχιστον και να υπάρχει και ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων από κάθε κράτος μέλος. τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη ε, και την αναλογία των Ευρωβουλευτών. Σημαντικά μέτρα είναι όλα αυτά για την πρωτοβουλία πολιτών, ε, για να έχει και κάποιο κύρος η πρωτοβουλία, για να, μην να θεωρείται έτσι σοβαρή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την πρωτοβουλία των πολιτών, είναι γεγονός ε, ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, καλή είναι η ενθάρρυνση των ε, πολιτών στη συμμετοχή, στη, στα ευρωπαϊκά δρόμενα κατόπιν υπογραφέ, ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Πάρα πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία, αλλά πώς θα την υλοποιήσουμε στην πράξη. Πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν ε, στις, ε, στη δημοκρατία μέσω των εκλογών. Και ίσως ε, θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτό να ενισχύσουμε την συμμετοχή των πολιτών. Βεβαίως η πρωτοβουλία των πολιτών είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει τον ενεργό ρόλο των πολιτών. Όμως ο κίνδυνος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην συνεχίσει την πρωτοβουλία αυτή. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συμπληρώσω και εγώ κάτι ε, για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι πολύ σημαντική, είναι ένα νέο πείραμα, την υποστηρίζουμε κι εμείς και θα πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή στην πράξη. Τώρα προβλέπεται μια τριετία όπου πραγματικά χρειάζεται μεγάλη παρακολούθηση για να δούμε αν είναι πραγματική πρωτοβουλία των πολιτών και να μην την καταχραστούν ας πούμε άλλα συμφέροντα ε, να είναι πραγματικά πρωτοβουλίες των πολιτών των ίδιων και όχι κάποιων άλλων ενδιαφερομένων. Και ελπίζω και εγώ προσωπικά να καταθέτουν οι πολίτες επικοδομητικές προτάσεις τραμμένες προς το μέλλον και να μην ε, το χρησιμοποιήσουν μόνο από την ε, αρνητική πλευρά. Με ιδιαίτερη προσοχή ακολούθησα την, παρακολούθησα την νομοθετική διαδικασία για την πρωτοβουλία των πολιτών και είμαι ικανοποιημένη ακόμα και με τις προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Επίσης, είμαι ιδιαίτερη περήφανη που μπορώ να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι στην Ιταλία μετά την έγκριση της οδηγίας για τα δοκιμές στα ζώα υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες και ενώσεις πολιτών που έχουν ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζονται μια πρόταση που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια πρόταση που θα οδηγήσει σε μια νέα νομοθεσία και που θα καταδικάζει τις δοκιμές που γίνονται στα ζώα. Πρόκειται για μια επιστημονικά μη αποτελεσματική μέθοδο και ιδιαίτερα επαχθή για τα ζώα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να υποβληθούν και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν, θα έχουν στόχο κοινοτικές αρχές. Uh, Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η πρωτοβουλία των πολιτών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες ε, να μιλήσουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προτάσεις που δεν της αρέσουν γιατί νομίζω μπορούμε να περιμένουμε πολλές πρωτοβουλίες που θα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερα, θα, θα τη ζητήσουν να είναι περισσότερο Ευρώπη και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, με ενθουσιασμό θα ανταποκριθεί, αλλά πώς ε, θα αντιδράσει σε προτάσεις για λιγότερη Ευρώπη ή σε προτάσεις για να γίνονται ορισμένα πράγματα καλύτερα, για μικρότερες δαπάνες ή για δηλώσεις κατά της ευρωπαϊκής φορολογίας. Πώς γίνει, πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις αυτές, ε, θα τις αντιμετωπίσει με σεβασμό, γιατί αν ανταποκρίνεται μόνο σε πρωτοβουλίες που ε, τις αρέσουν, τότε δεν έχει νόημα. Ένα ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπερψήφισα τις συστάσεις και τα σχετικά ψηφίσματα και πιστεύω ότι ο εισηγητή έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία και για μα και για τους πολίτες. Επίσης, εγκρίναμε τη συνθήκη της Λισαβόνας πρόσφατα στην Ιρλανδία, φαινόταν όμως για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι τα πράγματα θα περιπλέκονταν πολύ. Καταφέραμε, χάρη στην πρωτοβουλία των εισηγητών αυτή, να επιφέρουμε μία απλούστευση και έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο και το πάνελ των 7 μελών από 7 διαφορετικές χώρες. Πιστεύω ότι τα νέα αυτά μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι ανησυχίε των Ευρωπαίων πολιτών μπορούν να ληφθούν υπόψη και Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ε, στην Ιρλανδία λέμε ότι ε, μια καλή αρχή είναι ήδη το ίμιση της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Τι να σας πω, ε, δεν θέλατε να ακούσατε του Ευρωπαίου πολίτε πριν από την ε, έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα Για να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Φόξ προηγουμένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν αξίζει τον κόπο μια πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί δεν έχει καμία δεσμευτική, ε, δεν δεσμεύεται, μπορεί να παραγνωρίσει εντελω μια πρωτοβουλία και βλέπουμε και πάλι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν λαμβάνει υπόψη τι των Ευρωπαίων Ευρωπαίων πολιτών. Παρακαλώ πολύ, ακούστε επιτέλους Ευρωπαίους πολίτες. Περνάμε τώρα στην ε, παρουσία του προγράμματος της Εργασίας Επιτροπής για το 2011. Ο κύριος Higgins για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2011. Η χρηματοπιστωτική κρίση είναι η μεγάλη πρόκληση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσω και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στου στόχου που έθεσε. Όσον αφορά την, το ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό από απόψεω ε, κεραιότητα και συνοχή ε, τη Ευρωζώνη ε, και στο πλαίσιο τη αλληλεγγύη, επειδή υπάρχει ένα κοινό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προστατεύσουμε. Όσον αφορά την απασχόληση και την οικονομία, χαίρομαι ιδιαίτερα που τον Ιανουάριο του 2011 θα εγκρίνει την πρώτη ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη που θα αναλύσει την οικονομική κατάσταση τη ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ενδεχόμενε ανισορροπίες και συστημικούς κινδύνους. Αυτό νομίζω ότι είναι μια σωστή κίνηση προς την ευφυή οικονομία. Είμαστε μια κοινότητα 5,5 εκατομμυρίων ε, ανθρώπων. Ε, πρέπει να, να ενισχύσουμε τη θέση μα στην διεθνή πολιτική σκηνή και εύχομαι στην, στην Επιτροπή κάθε επιτυχία. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα. Ε, είναι πολλές οι παράγραφοι, αλλά η πιο περίεργη είναι αυτή που υποχρεώνει τα κράτη να δίνουν το 0,7% του ΕΕ στην αναπτυξιακή βοήθεια και να φροντίζει μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόζονται αυτά. Έχει νόημα αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια. Και είναι ε, βαριά παραβίαση αυτή ε, της αρχής επικουρικότητας. Και στην παράγραφο 52 καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκμεταλλευτεί, λέει, την ευκαιρία. Ε, ποια ευκαιρία τη διεύρυνση. Μα, το, επανειλημμένες προκλήσεις της Τουρκίας, μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξισλαμισμός προϊόν. Περνάμε τώρα στο μέλλον της στρατηγικής ε, σχέσης Αφρικής-Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ο κύριος Κλέης πάλι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα το ψήφισμα έχει αυτό ε, και καλά στοιχεία, όπως είναι η καταδίκαση ε, της συμμετοχής, η καταδίκη συγγνώμη, της συμμετοχής ε, του ε, εγκληματία Μπουγκάμπη στη Σύνοδο Κορυφής Λισαβόνας, που είναι και φυγάς κατά τα άλλα. Επίσης, υποστήριξη της Γεωργίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την άλλη όμως, και πάλι πρέπει να ξεφορτωθούμε το ανόητο 0,7%. 60 χρόνια έχουμε στείλει ένα δισεκατομμύριο δολάρια στην Αφρική και τι ε, προκαλέσαμε μεγαλύτερη εξαχθλίωση. Αν χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια ε, θα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε την παράνομη διαφυγή κεφαλαίου. Σωστά επίσης στιγματίζει το ψήφισμα. Και καταψήφισα γιατί για τη μετανάστευση αυτά που λένε τα χειρότερα. Ε, ο κύριος ε, Καμάλ, για ένα λεπτό. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν βλέπουμε την δινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πάρα πολλές χώρες αφρικής, Αφρική, λέμε ότι σαφώς θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιμέρου κάτω τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσουμε να βγουν από τη φτώχεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όμως πιο αποτελεσματικοί. Κάθε φορά που υπάρχει μια καταστροφή, Σαφώ η βοήθεια θα πρέπει να παίζει βραχυπρόθεσμα ένα σημαντικό ρόλο. Μακροπρόθεσμα όμω πολλέ φορέ δεν κατανέμεται σωστά η βοήθεια που δίνουμε. Και αυτό δεν είναι σωστό για του φορολογούμενου σε διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστέλουν χρήματα σε κυβερνήσει στην Αφρική, οι οποίε δεν διακυβερνούν σωστά την ε, χώρα τους και που δεν δίνουν σωστά τα χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη είναι να βοηθήσουμε του επιχειρηματίες στις φτωχές χώρες. Αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο στις δικές τους κοινότητες και μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να βγάλουν τους δικούς τους ανθρώπους από τη φτώχεια. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις αγορές μας και ας στοχεύουμε περισσότερο την βοήθεια που στέλνουμε προς την ανάπτυξη πραγματικά και την εξάλληψη τη φτώχειας. Ευχαριστώ. Ο Χάναν για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαζί με πολλούς συναδέλφους πήγα στη Σύνοδο ΑΚΕ στην Κινσάσα που ήταν ε, ε, η δεύτερη χειρότερη χώρα βέβαια στον κόσμο. Ε, είναι πάνω από τη Ζιμπάμπουε. Όμως οι Κογκολέζοι δεν μπορούν να πούν στον εαυτό τους ότι πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση για να αλλάξει η κατάστασή τους. Η, δημοκρατία του Κονγκό, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ε, υπερβάλλει στην τραγική κατάσταση της Αφρικής. Ενδεχομένως η επικιοκρατία να, ε, είναι πιο εύκολο να την κατηγορήσει κανείς από ε, τις γειτονικές χώρες. Υπάρχει βέβαια και η κατάρα των φυσικών πόρων που κόβει το δεσμό μεταξύ της διαφθοράς και των πολιτικών. Υπάρχει επίσης και η έλλειψη ταυτότητας ε, εθνικής ή γλωσσικής ταυτότητας. Ε, ε, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε ότι ο πατριωτισμός οδηγεί σε πόλεμο. Εγώ θα ήθελα να σας δείξω ότι μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό καταφέρατε να περάσετε το χρόνο. Συνήθως ε, είστε, σέβεστε το χρόνο σας, αλλά αυτό είναι ένα ρεκόρ στην προσωπική σας ε, ιστορία. Θα ήθελα όμως ε, να σας συγχαρώ για τις υπόλοιπες φορές που έχετε σεβαστεί το χρόνο. Τροπίζει το 2011 ο κύριος Σέια. Thank you very Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, χώρες ε, οι οποίες έχουν βρεθεί σε ευνοϊκότερη κάπως θέση. Προσπαθούν να προσελκύσουν περισσότερους πόρους. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτερε πάντω, τρει μεγαλύτερε πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξαν τα όσα λέγονται στο κείμενο για τα ταμεία αυτά. Και πιστεύουμε επίση ότι ο πρώτο πυλώνα θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Η Ουγγαρία χθε έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα εγκρίνοντα ένα σχετικό τέτοιο νόμο. Επίσης, η όλη συζήτηση για τις λευκές και πράσινες βίβλους θα πρέπει να γίνεται στο ίδιο πνεύμα. Πρόεδρε, η νέα θεσμική αρχιτεκτονική που προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνας τονίζει ότι η προστασία και προώθηση των θεμελιδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η δημοκρατία και το κράτο δικαίου στην Ευρώπη και η βάση για αυτά. Εγώ υποστήριξα την έκθεση γιατί ε, θεωρώ ότι χρειάζεται νέος ορισμός ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο ιστορικό της Ένωσης, αποτελεσματικός και οργανικός, να υπάρχει ευθύνη και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί καθημερινά διαπιστώνουμε παραβιάσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πούμε ότι έχει αλλάξει ε, άρδιν ε, η νομική κατάσταση στην Ευρώπη ε, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας και χρειάζεται εξυγχρονισμός και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικά, οικονομικά, αλληλεγγύη και τα δικαιώματα της τρίτης γενεάς. Ο κύριος Αντινόρο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αποφάσισα να υπερψηφίσω την έκθεση αυτή γιατί όχι μόνο επειδή το ζήτησε αυτό η πολιτική μου ομάδα, αλλά επειδή είμαι πεπισμένο ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί Σαφώ έχουμε νέε αρμοδιότητε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά διαρθρώνονται όλο και καλύτερα οι αρμοδιότητε αυτέ. Το είδαμε επίση αυτό και με την σημερινή ψηφοφορία που έγινε για τον προπολογισμό. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια κοινή θέση σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκθεση αυτή. Καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό μέσω των συμβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εξαιρετική εργασία που έχει κάνει η Κίνγκα Γκάλ και πιστεύω ότι με την έκθεση αυτή θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τη δραστηριότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εδώ. Ο κύριος Στάκουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Κίνγκα Γκάλ για μια εξαιρετική έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω είναι μόνο μία έκθεση αυτή. Δεν πρέπει να μα διαφεύγει ότι έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά στην πράξη. Για παράδειγμα, μεγάλε μειονότητε Ρωμά ε, είναι μια περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίση, η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Μόλις απονείμαμε το βραβείο Ζαχάροφ. Όμω υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλλειψη ελευθερίας ε, έκφρασης. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να φρουρούνται γιατί ε, φοβούνται για τη ζωή τους όταν εκφράζουν τις απόψεις τους. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές φορές ακόμα και στα πλαίσια του ίδιου του Ιταλικού κράτους βλέπουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το βλέπουμε αυτό στη Συμφωνία Ιταλία-Λιβύη αλλά επίση και στο νομοσχέδιο Μπαβάλα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υποστηρίζεται από ένα κοινοβούλιο με τρόπο όμως αντιδημοκρατικό. Οι πολίτες δεν μπορούν να εκφράσουν μια συγκεκριμένη υποστήριξη. Χθες είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Είδαμε επίσης πώς ψήφισαν συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ πολύ, μιλάμε λοιπόν για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν γίνει ακόμα και κάποιες καταγγελίες για ε, διαφθορά όσον αφορά τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι υπερψήφισαν την κυβέρνηση Μπερδουσκόνη χθες. Θα δείτε επίσης κάποιες αποφάσεις ε, των ε, Ιταλικών ε, δικαστηρίων. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε έτσι, δεν, έχετε, δεν σας έχω δώσει το λόγο και δεν μπορείτε να αποσπάτε έτσι τους υπόλοιπους ομιλητές. Παρακαλώ, συνεχίστε, σας δίνω ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Στι Στις 9 eh, Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την ημέρα κατά της διαφθοράς. Χθες το Ιταλικό Κοινοβούλιο ε, ενέκρινε, αν θέλετε, την πρώτη μέρα υπέρ της διαφθοράς των βουλευτών του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Do you, would you... Είναι η τελευταία φορά που σας το λέω. Εσείς εκεί στο βάθος. Αν σηκωθείτε και πάλι και διακόψετε τη συνεδρίαση θα σας ζητήσω να αποχωρήσετε. Σας είναι σαφές. Παρακαλώ μην το ξανακάνετε. Τελειώσατε. κύρια ε, Κύριε Αλφάνη, θέλετε ακόμη χρόνο. La Presidenza ha sentito, i colleghi hanno sentito l'intervento, io avrei... Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι με άκουσαν. Αν δεν με άκουσαν κάποιοι συνάδελφοι μπορώ να ξαναπώ τα όσα θέλω να πω. No, Mr. Eh, Mrs. Pietikainen, if she's not here, she's here. Yes, she's here, okay. Κυρία Πιετικάιν, είναι εδώ. Arvoisa puhemies, ε, Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας, κάποιες, ε, κάποιοι βασικοί τομείς ε, ευημερίας ε, των ε, πολιτών έχουν συμπεριληφθεί στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρέπει να επικεντρωθούμε στην, στον έλεγχο του σεβασμού των ανθρωπίνων αυτών δικαιωμάτων ε, και να τα προωθούμε σε όλους τους τομείς πολιτικής, σε όλα τα κράτη-μέλη, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. Είναι σημαντικό όλοι να δουλέψουμε προς αυτό το κοινό στόχο. ώστε ό,τι ε, μπλοκάρεται στο Συμβούλιο να μπορεί να προχωρήσει και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε κάθε φορά που υπάρχει παράβαση των ε, θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Yeah, thank you. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε είναι αυτονόητο ότι καταψήφισα αυτή την πολιτικός ορθή έκθεση. Ως ε, φλαμανδός δημοσιογράφος θεωρώ απαράδεκτο ότι το Κοινοβούλιο ε, εξισώνει τον εθνικισμό με ε, τη διάκριση και την ξενοφοβία. Και καλούν, λέει, να προσφύγουμε κατά των κρατών μέχρι να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν χρειαστεί επίσημη προσφυγή στο δικαστήριο για να παγώνουν κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή τα κράτη-μέλη τα θέτουμε υποκυδαιμονία, έτσι, απαράδεκτα πράγματα. Ε, μια πραγματική πολιτική ε, ε, απελάσεων στο μέλλον θα μπλοκάρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ξεφεύγει από τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κλασική αρμοδιότητα κράτου μέλους και όχι της Επιτροπής. Και τέλος ο κύριος Χάνεν μετά από μερικές λάθος ε, ε, σε μια παράγραφο ε, έχουμε δει ήδη από το παρελθόν ήδη από το 1984 του Όργολ για πώς μπορεί να διαστρεβλωθεί η ε, γλώσσα και η ε, ελεύθερη έκφραση. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Τι θα πει ελευθερία. Παλιά ήταν ελευθερία της λατρείας, της έκφρασης και τα λοιπά. Και τώρα ελευθερία σημαίνει δικαίωμα. Έχω ελευθερία να δουλεύω, έχω ελευθερία να είμαι ασφαλισμένο στο σύστημα υγείας. Αυτή η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ξεφύγει από την έννοια του δικαιώματος που είναι ως εγγύηση ανθρώπινης προσωπικής ελευθερίας σε ένα δικαίωμα που είναι αξίωση έναντι πάντων. Ότι έχω το δικαίωμα ε, να με ε, μεταχειρίζονται ίσα, αλλά τώρα έχουμε πλέον δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί. Ε, και αυτό έχει ξεφύγει από τους εκλεγμένους προσώπους του λαού σε μη εκλεγμένους. Ε, η κυρία Ροντσούλη, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σα ζητώ συγγνώμη για πριν, αλλά δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να δεχτώ κάτι τέτοιο. Και λυπάμαι που η κυρία Αλφάνο χρησιμοποιεί τι επεξηγήσει ψήφων για να μιλήσει για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην ιστορική πολιτική τη Ιταλία. Χθε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε υπέρ τη κυβέρνηση Μπερλουσκόνη με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Ε, Επομένω, θα ήθελα απλώ να σα πω και εγώ ότι ψήφισα υπέρ τη ε, έκθεση Γιουβάν. για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο που μπορεί να δραματίσει η διαφήμιση για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα στους Ευρωπαίου πολίτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θέλει να επιφέρει πιο συγκεκριμένους κανόνες σε έναν τομέα ο οποίος ε, φαίνεται να είναι όλο και πιο όριστος αυτή τη στιγμή και αφηρημένος, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία. Ξέρετε ότι πολλές φορές στα πλαίσια της τεχνολογίας αυτής μετακινούνται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ με την έκθεση Γιουβάν γιατί ακριβώς επικεντρώνεται και στις πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά τα οποία δέχονται όλο και περισσότερο πιο επιθετική διαφήμιση. Είναι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαφήμιση συχνά είναι χρήσιμη πληροφόρηση των καταναλωτών έτσι ώστε να καταναλώνουν και να επιλέγουν με τα λόγου γνώσεως. Υπάρχουν και κανόνες συμπεριφοράς και διοντολογίας στην, στη διαφήμιση. Αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα βέβαια. Έχει ε, εκφυλιστεί ε, αυτό και πολύ συχνά η διαφήμιση απευθύνεται σε παιδιά. Και ε, καλά κάνει το κοινοβούλιο και εκφέρει γνώμη γι' αυτό. Θα πρέπει να δοθεί και συνέχεια. Είναι ένα σημαντικό τμήμα η διαφήμιση τη εσωτερική αγορά για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και να, δώσουμε, να δοθούν επιλογέ στου καταναλωτέ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση γιατί δεν προτείνουμε νέα νομοθεσία, ούτε ρυθμίζουμε τη διαφήμιση, ούτε ελέγχουμε και περιορίζουμε το διαδίκτυο. Θέλουμε να αυξήσουμε την ευαισθησία για την ευθύνη των ε, διαφημιστών, όπως επίσης ε, και τις αθέμητες πολιτικές που χρησιμοποιούν σε σχέση με την ε, ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων. Ζητώ από την επιχειρηματική κοινότητα να αυτορυθμιστεί εθελοντικά να συμμετέχει σε προγράμματα προκειμένου να ε, μην ε, υπάρχει ε, υπερβολική διαφήμιση και ειδικότερα θα ήθελα να μην χρησιμοποιείται ο Batman, ο Spiderman εναντίον των παιδιών μας. Ευχαριστώ. Τέλος, η έκθεση Μπένστεν. Κύριος Higgins, για ένα λεπτό. one minute. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση αυτή, την υπερψήφισα. Θα πρέπει να εξοικονομούμε την ε, ενέργεια, ε, να μειώνουμε τη χρήση της και να έχουμε τελικά ενεργειακή απόδοση στην Ένωση. Πολύ συχνά ε, συζητούμε για τις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ξεχνούμε έτσι την κατανάλωση ηλεκτρισμού. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ρόντο, για ένα λεπτό. Thank you, Mr. President. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενδιαφέρον αυτό το οποίο με εσάς τους Ιταλούς συναδέλφους. Την προηγούμενη εβδομάδα πάρα πολλοί πήγανε στο Κανκούν Παρόλα αυτά όμως δεν έδωσαν την απαραίτητη μάχη για τις κλιματικές αλλαγές. Με τη σημερινή ψηφοφορία για την ενεργειακή απόδοση πιστεύω όμως ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά. Όπως λέει πολύ σωστά η έκθεση αυτή, η ενεργειακή απόδοση είναι ο πιο αποτελεσματικό γρήγορο τρόπο για να μειωθούν οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ουσιαστικά όμω τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη υστερούν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι με τι προσπάθειε αυτέ θα καταφέρουμε να πετύχουμε μόνο του μισού στόχου μα για το 20%. 20%. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση αυτή περιέχει πολλέ λύσει, οι οποίε όμω πρέπει τώρα να εφαρμοστούν στην πράξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπένσεν και να τον συγχαρώ για την εξαιρετική εργασία που έκανε για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Νάιτε για ένα λεπτό. Okay. Uh... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω ε, την έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντική ε, και σημαντική όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και μετά τα όσα συνέβησαν στην Κανκούν βρέθηκαν κάποιες λύσεις και θα πρέπει τώρα εμείς να τις εφαρμόσουμε, να τις ε, υλοποιήσουμε στην Ευρώπη. Η ενεργειακή απόδοση είναι από τις σημαντικότερες οδούς και τις πιο σωστές που έχουν επιλέξει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να καταρτήσουν τώρα εθνικά σχέδια ε, για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα και υποστήριξη βέβαια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους τομείς, για τις μεταφορές, για τις ε, κατοικίες, για την οικοδομή κτλ. Το έγγραφο αυτό είναι πολύ ωραίο για την οικονομία μας. Arvoisa puhemies, minä myös äänestin tämän Pentsenin energiatehokkuutta Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα και εγώ την έκθεση Μπέντσεν για την ενεργειακή απόδοση. Στην Ευρώπη έχουμε δεσμευτεί να ε, κάνουμε οικονομία ενέργειας και να ε, βρούμε νέες ε, μορφές κατανάλωσης ενέργειας. Όταν ορίζουμε αυτούς τους στόχους όμως, θα πρέπει όλοι να αισθάνονται την ίδια δέσμευση και την ίδια ευθύνη και την ίδια προσήλωση. Ωραία είναι οι στόχοι και τα ευχολόγια, αλλά κανένας δεν τους έχει χωνέψει ακόμα. Και αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την Ευρώπη, αλλά ε, και τον κόσμο όλο. Δεν θα πρέπει να βάζουμε εμείς εμπόδια στην ανταγωνιστικότητά μας, αλλά ε, να είμαστε παγκόσμια αγωνιστικοί και να παραμένουμε. Κυρία Αλφάνο, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πιστοδρομήσει στην πρόκληση για την ενέργεια που απασχολεί όλο τον πλανήτη. Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας δεν θα πρέπει να συνδέεται αναγκαστικά με την ενεργειακή της κατανάλωση. Η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους, λιγότερη ενέργεια και να έχει και μεγαλύτερη παραγωγικότητα παράλληλα. Επίσης, δεν θα πρέπει να, κατα... να βασίζεται η οικονομική ανάπτυξη μόνο στην ε, μεγαλύτερη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Επομένως, η ενεργειακή απόδοση πιστεύω ότι αποτελεί πραγματικά πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπης στο οικονομικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει τους, ε, τις απαραίτητες αποφάσεις και να ακολουθήσει ουσιαστικά τους στόχους που έχει θέσει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα και εγώ την έκθεση αυτή. Είναι φιλόδοξη και ζητώ και είναι και δεσμευτική η γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Χαίρομαι ε, με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή μόνο με διεθνείς ε, στόχους και συμφωνίες. Χρειάζονται και πρακτικά μέτρα συγκεκριμένα για να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας απόδοση και για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο χρειάζεται συνολική προσέγγιση αλλά πάντα δεσμευτική γραμμή με κυρώσεις τελικά εφόσον θα είναι δεσμευτική. Πολύ καλό το πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος... Ε, are you, are you applauding me or you ask, you... Με χειροκροτάτε ή ζητείτε διαδικαστικό στι επεξηγήσει ψήφου που είναι περίεργο να το κάνει κανεί, αλλά έχετε το λόγο. E Θα ήθελα να θέσω ένα διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο δέχεστε αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιείτε ο χρόνος από τις επεξηγήσει ψήφου για να δίνετε δυνατότητα σε κάποιους συναδέλφου να προσβάλλουν τελικά τους ίδιου Ιταλούς, την Ιταλική κυβέρνηση, τη στιγμή που η Συνάδελφο μίλησε ε, κατά τη Ιταλικής κυβέρνησης, τη στιγμή που οι εθνικοί βουλευτές ε, ενέκριναν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο την ε, κυβέρνηση Μπερλουσκόνη νομίζω ότι δεν θα πρέπει σύμφωνα με τον κανονισμό να γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί διαφορετικά σε όλε τι μελλοντικέ επεξηγήσει ψήφου θα παίρνω και εγώ το λόγο για να μιλήσω υπέρ τη κυβέρνηση αυτή η οποία νόμιμα έχει την εξουσία με την υποστήριξη του τελικού κοινοβουλίου. Ελπίζω να εκτιμάτε το γεγονό ε, ότι σα έδωσα το λόγο παρά το γεγονό αυτό που είπατε δεν είναι διαδικαστικό η δουλειά μου δεν είναι να παρακολουθώ τι θέλουν να πούν ε, οι βουλευτές. Η δουλειά μου είναι να εξασφαλίζω ότι το λένε όταν έχουν το λόγο ε, για να το πούν, αντί να διακόπτουν ένα τον άλλον και μάλιστα με έναν ε, αρκετά δυνατό, ηχηρό και αγενή τρόπο. Θα ήθελα να ζητήσω να είστε πολιτισμένοι ο ένας προς τον άλλον και παρακαλώ και προσπαθώ επίσης να κρατάω και το χρόνο αυτό που λέγεται σε, μια δημοκρατική, ένα δημοκρατικό όργανο είναι η δική τους δουλειά και όχι η δική μου. Και έλεγε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μερικά ε, σημεία θα ήθελα να θέσω για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι τώρα έχουμε προσέξει πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντικές αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και γι' αυτό ακριβώς χαιρετίζω αυτήν την έκθεση. Ειδικότερα σε σχέση με τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, ακόμη και αυτό το κτίριο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, Μιλάνε πίσω μου και δεν ε, μου επιτρέπεται να συνεχίσω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, συνεχίζω. Στον τομέα λοιπόν των κτηρίων θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα και ειδικότερα σε σχέση με το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και το ε, κτίριο των Βρυξελών. Ε, είναι πολύ σημαντικά και θα έπρεπε να είναι ενεργειακώ πιο αποδοτικά. Ένα ακόμη είναι το θέμα των μεταφορών. Ε, Μηχανέ δίζελ θα έπρεπε να είναι πιο αποδοτικέ και οι κατασκευαστέ θα έπρεπε να τι κάνουν πιο αποδοτικέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, δουλειά της πράσινης ε, σημαίας. Οι διευκρινήσεις ψήφου ε, διακόπτει τη συνεδρίαση ως τις 3 το απόγευμα. Thank you so much.